Ακολουθεί η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ερώτηση του κυρίου Σάρλα Γκέρενς, εξ ονόματος της Ομάδας των Φιλελευθέρων, με θέμα το πρόβλημα της περιορισμένης πρόσβασης των υποανάπτυξη χωρών σε ορισμένα εμβόλια. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς, συντάκτης ερώτησης, για δυόμιση λεπτά. Σάρλ, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντός του πλαισίου της ε, ερώτησης αυτής προς την Κομισιόν, θα ήθελα να εξερευνήσω τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σταματήσει μια διαδικασία που εμποδίζει τα 90% του πληθυσμού να έχουν πρόσβαση στα εμβόλια για τη γρήπη ή τα 1 ή 1. Και γενικά την πρόσβαση στα εμβόλια. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινοφανέ. Πράγματι, το πρόβλημα αυτό τίθεται κάθε χρόνο σε σχέση με την εποχική γρήπη. Εν γέννη, οι νέοι ιοί της εποχικής γρήπη εμφανίζονται καταρχήν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και από τη στιγμή εκείνη, τα εργαστήρια, τα φαρμακευτικά των αναπτυγμένων χωρών ξεκινούν τη διαδικασία παραγωγής εμβολίων και χρειάζεται να έχουν στελέχη τα οποία προέρχονται κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες αυτές μορφές ιών. Από τη στιγμή που τελειοποιούνται τα, τα εμβόλια μπορούν να προστατεύσουν απλώς και μόνο τον πληθυσμό των αναπτυγμένων χωρών ενώ οι πληθυσμοί των χωρών του Νότου μένουν ανυπεράσπιστοι ενώπιον της πανδημίας. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν τι θα κάνει για να σταματήσει αυτή η αδικία. Είναι ηθικά υπερασπίσιμο να δίνουμε προστασία μονάχα σε ένα τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν το απαραίτητο βαλάντιο. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε κατά πόσο η Κομισιόν θέλει να μας αναφέρει ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβει για να μπορέσει να καλύψει αυτό το κενό. Και ποια θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως η στατιστική, στρατηγική συγγνώμη της Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη και με τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών ή ακόμα και με συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για να υπάρξει μια διαδικασία που θα επιτρέψει στους κατοίκους των αναπτυσσομένων χωρών να έχουν πλήρη πρόσβαση στα εμβόλια. Το καθεστώς του ΠΟΕ για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί πράγματι ένα εμπόδιο για την παραγωγή εμβολίων από τις αναπτυσσόμενες χώρες ή όχι, ρωτώ την Κομισιόν. Εάν ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ξεκινήσει μια συζήτηση στα πλαίσια του ΠΟΕ με στόχο την εξάλληψη ρητρών αυτού του είδους. Και ένα τελευταίο ερώτημα προς την Κομισιόν. Μπορεί η Κομισιόν θα, να μας αναφέρει ποια μέτρα θα λάβει για να βελτιώσει το επίπεδο των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι απαραίτητο στοιχείο μιας πιο ισοδίκαιας πρόσβασης στους εμβολιασμούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ φίλε Γκέρενς δίνω το λόγο στον φίλο επίτροπο Όρμπαν για να απαντήσει εξ ονόματος της Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκιόρενς για το ερώτημα το οποίο έθεσε. Με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης μπορώ να αναφερθώ τόσο στα θέματα τα οποία άπτονται άμεσα της ε, πανδημίας γρήπης ή τα 1 1, αλλά μπορώ να αναφερθώ και σε άλλες πτυχές των ενεργειών της Κομισιόν με στόχο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που επικρατεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δράσει ταχαίως τόσο στο εσωτερικό της και όσο και στο εξωτερικό της σε σχέση με την πανδημία αυτή. Πράγματι, Πρόκειται για μια κρίση η οποία αποτελεί, απαιτεί μια συνολική, μια παγκόσμια προσέγγιση. Όχι μόνο για λόγους αποτελεσματικής προστασίας των πολιτών μας, αλλά επίσης για να εκφράσουμε και την απαραίτητή μας αλληλεγγύη προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αναφερόμαστε στο θέμα της ε, αποτελεσματικότητας, γιατί το σύστημα της πρόορης προειδοποίησης για να αντιμετωπίσουμε την ταχαία εξέλιξη της πανδημίας, είναι απαραίτητο να μας οδηγήσει σε ταχεία λήψη μέτρων στις χώρες όπου έχει εμφανιστεί ήδη η πανδημία. Όλα αυτά είναι απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε τη στρατηγική μας και να την προσαρμόσουμε στις υφιστάμενες συνθήκες. Αλλά μιλάμε επίσης και για το θέμα της αλληλεγγύης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κυριότερος χορηγός προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και ως ε, προνομιακός εταίρος ενός μεγάλου αριθμού αναπτυσσομένων χωρών είναι υποχρεωμένη να σταθεί στο πλευρό των χωρών αυτών να τις βοηθήσει για να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα απειλή. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει από συγκεκριμένες αρχές. Δεν ξεκινάει από το μηδέν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εμπειρία μας με τον ιό ΙΤΑ 5 νη 1 μας επέτρεψε με την ε, συνεργασία της Παγκόσμιας Τράπεζας του ΠΟΕ μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικές διαδικασίες για να μπορέσουμε να συντονίσουμε την τεχνική αρρωγή, να δώσουμε την απαραίτητη πληροφόρηση στον πληθυσμό και να ξεκινήσουμε ορισμένα εργαλεία χρηματοδοτικού χαρακτήρα, παραδείγματος ένα ειδικό ταμείο στα πλαίσια της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως είπε και η κυρία Τσάνγκ, η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, του ΠΟΗ, συγγνώμη, του ΠΟΕ, ο κόσμος βρίσκεται ενώπιον μιας πανδημίας η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια του συστήματος αντιμετώπισης αυτών των υγειονομικών απειλών. Υπάρχουν στοιχεία αυτής της απειλής που θα τα επεκτείνουμε σε άλλες μορφές γρήπης και σε άλλες ενδεχόμενες πανδημίες. Προφανώ είναι απαραίτητο να ευνοήσουμε τον εμβολιασμό στι αναπτυσσόμενε χώρε. Έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και έχουμε ξεκινήσει ακόμα και μία συζήτηση εδώ και δύο χρόνια μέσα στα πλαίσια του ΠΟΥ και στην ομάδα εργασία που είναι ειδική για τι πανδημίε. Ο ΠΟΥ λοιπόν είχε την ιδέα να δημιουργήσει αυτή την ομάδα εργασία. Και αυτή τη βδομάδα στην Γενέβη, ο ΠΟΗ θα παρουσιάσει τα πρώτα πορίσματα αυτής της ομάδας εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέσχει με τρόπο ιδιαίτερα ενεργό στις εργασίες Τα τελικά πορίσματα και οι συστάσεις θα παρουσιαστούν στο Εκτεριστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα λάβει χώρα στο τέλος Ιανουαρίου. Από τότε, από το έκτοτε, θα γνωρίσουμε λοιπόν ποια θα είναι η καλύτερη ισορροπία μεταξύ αφενός των κινήτρων προς την έρευνα και την ανάπτυξη για να αναπτυχθούν νέα φαρμακευτικά σκευάσματα και αυτό βέβαια αφορά περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα γιατί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τους ιούς είναι σημαντικά και θα πρέπει να δοθεί λοιπόν αυτή η παρότρινση προ τι φαρμακευτικέ εταιρείε. Επίση όμω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισοδίκαια πρόσβαση στα προϊόντα τα οποία θα προκύψουν από αυτή την έρευνα καθώ και την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιε επιφυλάξει έναντι οποιασδήποτε προσπάθεια να περιοριστεί η χρήση βιολογικού υλικού για να μπορέσει να γίνει η απαραίτητη έρευνα στον τομέα αυτό. Η ενεργή λοιπόν συνεργασία σε διεθνέ επίπεδο με τρόπο διάφανο και κάτω από την υποστήριξη φορέων όπως είναι ο ΠΟΗ είναι κάτι το οποίο είναι απαράγραπτο και να μπορέσουμε εμείς να διανύμουμε με ταχύ ρυθμό τους τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη μαδημία ή τα ένα ή ένα. Αυτή η νέα πανδημία λοιπόν, για την οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν εμβόλια, αντιμετώπισε προβλήματα παραγωγικής ικανότητος διότι υπήρξαν μαζικές αιτήσει από τις χώρες που έχουν τις ε, ικανότητες να αγοράσουν τέτοια εμβόλια. Ορισμένοι παραγωγοί εμβολίων και ορισμένε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να ε, σχηματίσουν αποθέματα σε ύψος 10% των αναγκών τους για να μπορέσουν να βοηθήσουν δωρεάν ή σε χαμηλή τιμή χώρες οι οποίες αναπτυσσόμενες. Αυτό μας δίνει την εντύπωση και την ελπίδα ότι υπάρχει πράγματι αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Κομισιόν η βοήθεια προς τις τρίτες χώρες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πανδημία είναι κάτι το οποίο θεωρούμε απαραίτητο και δεν θέλουμε να περιοριστούμε μονάχα στα, στο θέμα των εμβολίων από τη στιγμή που τα εμβόλια αυτά θα είναι διαθέσιμα. Είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε και να εδραιώσουμε τα υγειονομικά συστήματα των χωρών αυτών. Αυτό είναι μια βοήθεια που δίδει η Κομισιόν και τα κρατημέλη με πολλούς τρόπους, αρρωγή σε συγκεκριμένα σχέδια, υποστήριξη στον προϋπολογισμό των χωρών αυτών που είναι ε, εταίρες μας και γενικά υποστήριξη προς τους διεθνείς οργανισμούς. Πρέπει οι χώρες, οι αναπτυσσόμενες, να έχουν τα ενία της ίδιας τους της ανάπτυξης και πρέπει να δεσμευθούν και από τη δική τους πλευρά ώστε η αρρωγή που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αποτελεσματική. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε από πολύ κοντά το θέμα της εξέλιξης της παθολογίας των ιών αυτών για να καθορίσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία χρειάζεται να έχουμε καλύτερα εξοπλισμένα υγειονομικά συστήματα για τον εντοπισμό, για την έγκαιρη αντιμετώπιση και θεραπεία των περιστατικών και για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την ισότιμη ε, πρόληψη με τα απαραίτητα εργαλεία όταν αυτή είναι απαραίτητη. Σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει και να κινητοποιήσει και τα εργαλεία της έκτακτης ανθρωπιστικής υποστήριξης με τρόπο ο οποίος θα είναι εύκαμπτος για την χρησιμοποίηση ήδη υπαρχόντων μέσων τα οποία μας συνδέουν με τις χώρες αυτές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Εάν προκύψει κάποια σοβαρή απειλή σε υγειονομικό επίπεδο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο. Γνωρίζει δε η Κομισιόν ότι δύναται να βασίζεται στην αποτελεσματικότητα και την θέληση αυτών των φορέων. Ευχαριστούμε. Θα λάβουν το λόγο τώρα οι ομιλητές εξ ονόματος των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Πρώτος ο κύριος Γκέι Μίτσελ του ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν έρχεται πανδημία γρήπης, ε, η είδησή της ε, το φέρνει στο προσκήνιο αυτό. Το πρόβλημα είναι όμως μόνιμο και διαρκές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η σημερινή προφορική ερώτηση ε, δείχνει πολύ εύγλωτα ποια είναι η υποκρισία ε, του δυτικού κόσμου και των αναπτυγμένων χωρών που δεν αφήνουν τι αναπτυσσόμενες χώρες ε, να ε, προστατεύσουν τον πληθυσμό τους. Οι ίδιες προστατεύουν το δικό τους πληθυσμό και μετά το πουλάνε στις φτωχές χώρες. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα έτσι ώστε οι φτωχότεροι του κόσμου που είναι και πιο εκτεθειμένοι ε, στην ασθένεια να έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν αυτό που εμείς στη Δύση θεωρούμε δεδομένα. Δηλαδή να προστατεύονται από νόσους που προλαμβάνονται. Βλέπουμε την αντίφαση και αντίθεση που υπάρχει με τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ρουτίνα το εμβόλιο BCG ας πούμε, στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο, 80% αποτελεσματικότητα και τελικά ε, η φυματίωση ε, δεν είναι η απειλή που υπήρχε στο παρελθόν. Αντίθετα, το 26% ε, των θανάτων από νόσους που προλαμβάνονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο οφείλονται στη φυματίωση. Αυτό τι δείχνει ότι αερογενείς νόσοι υψηλή ε, μεταδοτικότητας που πολύ εύκολα μπορούν να μεταδοθούν ε, ε, είναι πολύ συχνές στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η μισή ασθενής από AIDS στην υποσαχάρια Αφρική θα προσβληθούν από φυματίωση και βλέπετε πόσο τυχεροί είμαστε, τυχεροί είμαστε εμείς που ζούμε σε ένα περιβάλλον σχετικά ανοσοποιημένο. Χρειάζεται γενικότερα αναπτυξιακή βοήθεια. Αρκεί να δει κανείς τι γίνεται με την παροτίτιδα ε, στην Αφρική. Από το 2000 έχει πέσει κατά 90% επιπολασμός. Από το 2000 μέχρι το 2006. Κύριε ε, Πρόεδρε, είναι σαφές ότι έχει αποτελέσμα το εμβολιασμός και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας απευθύνω επίγουσα έκκληση να διατηρήσουμε την πίεση που χρειάζεται. Και ένα διαδικαστικό πριν τελειώσω κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, κάντε κάτι για τους αελκυστήρε εδώ μέσα. Ανεβοκατέβαινα, ε, δεν μπόρεσα σχεδόν να φτάσω την ώρα μου, ήταν σε συμφόρηση τα σανσέρ, κάτι πρέπει να γίνει εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ. Σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σας, θέλω να σας αποκαλύψω ένα απόρριτο των συζητήσεων στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Στην τελευταία συνεδρίαση του Προεδρείου κατήγγυλα την κατάσταση που μόλις μας περιγράψατε και δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό μόνο στο Στρασβούργο αλλά και στις Βρυξέλλες. Είχαμε εβδομάδες όπου ήταν πραγματικά αδύνατο να κινηθεί κανείς μέσα στους διάφορους λαβύρινθους που είναι τα κτίρια μας, γιατί δεν δούλευαν τα σανσέ. Λοιπόν, ελπίζω να διαβιβάσουμε από το Προεδρείο στις αρμόδιες υπηρεσίες το θέμα αυτό για να βελτιωθεί με κάποιο τρόπο η υπηρεσία στο σανσέρ. Και τώρα ο κύριος Κάσμαν εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ε, ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε να φύγουμε λίγο από τις ανελκυστηρίες και να επιστρέψουμε στα εμβόλια που προλαμβάνουν θανάτους, διότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε. Και βέβαια υποστηρίζω την έκκληση για την ΙΤΑ 1 1 αλλά θα ήθελα να το διευρύνω λίγο. Και επίτροπε υπάρχουν συστήματα που λειτουργούν και τα εμβόλια υπάρχουν ε, βακτηριογενείς ε, λοιμώξεις με μηνυγκίτιδα πνευμονία και συψεμία και είναι άγνωστες αρρώστιες ενώ μπορούν να προληφθούν από εμβολιασμό παιδιών κάτω των 5 ετών. Πνευμονία ε, που κάνουν να χάνουν τα παιδιά τους 2 εκατομμύρια παιδιά το χρόνο. Και είναι παγκόσμια πρόκληση αυτή για την υγεία με λύσεις. Μπορεί να σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι η Κομισιόν και πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, κάνει ε, υποσχέσεις μέσω ενός διεθνούς μέσου για ανοσοποίηση του πληθυσμού για τον πνευμόνιο κοκό. Κάτι που δεν αναφέρατε εσείς στην ομιλία σας. Μπορούμε και φίλουμε να κάνουμε περισσότερα για να γίνει προτεραιότητα ο πνευμονιό κοκός και να συνεργαστούμε με τις αναπτυσσόμενες χώρες για να κάνουν και αυτές το ίδιο. Αυτή η αντιμετώπιση του πνευμονιοκόκου είναι ε, πρωτοφανής ευκαιρία για τις χώρες να προστατεύσουν τα παιδιά τους από αυτό το νόσημα που σκοτώνει αλλά προλαμβάνεται. Από τις 71 χώρες ε, που είναι επιλέξιμες, οι 20 ζήτησαν χρηματοδότηση ε, για αυτό το πρόγραμμα που θα σώσει τόσες πολλές ζωές. Θυμίζω στο σώμα ότι είναι μοχλός για την ανάπτυξη των στόχων της χιλιετίας η πρόσβαση στα εμβόλια. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά 2 τρίτα μέχρι το 2050. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα εμβόλια αυτά θα πάνε στις χώρες που το χρειάζονται περισσότερο. Είναι απλό το βήμα και απλούστατα μπορούμε να σώσουμε εκατομμύρια παιδιά. Υπάρχει γραπτή δήλωση για αυτό το θέμα εδώ στο Κοινοβούλιο και ε, επίσης ε, ε, γίνεται λόγο για τι ευρεσιτεχνίε και πώ αυτέ θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει εξ ονόματος των φιλελευθέρων η κυρία Φρεντερή Κρυ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τούτη εδώ τη εβδομάδα, τα κράτη-μέλη μας προχωρούν στο πρώτο κύμα εμβολιασμού κατά τη γρήπη Α, ενώ ταυτόχρονα αναγκαζόμαστε παράλληλα να διαπιστώσουμε πόσο λίγη πρόοδος έχει γίνει στην ίδια αυτή η ιστορία των αναπτυσσόμενων χωρών. Ακούσαμε ότι εκατομμύρια προσώπων και παιδιών πεθαίνουν κάθε χρόνο σε αυτές τις χώρες από διάφορες νόσους που ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφός μου Γκέι Μίτσελ. Δεν λέω ότι είναι απλή η λύση βέβαια διότι το θέμα της πρόσβασης στα εμβόλια δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμο με την πρόσβαση στα φάρμακα. Είναι περιορισμένη η παραγωγή, είναι δύσκολο να υπάρχει η αλυσίδα, η ψυχρή, τη ψήξη των εμβολίων. Και επίσης ε, ακούσαμε ότι έχουμε 3 δισεκατομμύρια δόσεις το χρόνο. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια παγκόσμια στρατηγική και επειδή δεν έχω και χρόνο, τελειώνω Πρόεδρε, ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την έκκληση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για διανομή ε, εμβολίων, ιδιαίτερα εκεί που έχουμε μεγάλη φνησιμότητα, να Έχουμε και ΣΔΙΤ, συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για να καταπολεμήσουμε αυτή την έλλειψη εμβολίων. Ευχαριστώ. Και εξ ονόματος τώρα της ομάδας της Ενωτικής Αριστεράς, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ θέλω να τονίσω τη σημασία του ερωτήματος του κύριου Γκέρενς, γιατί είναι από τα πιο βασικά θέματα δικαιοσύνης. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση της πανδημίας της ε, γρήπης ΙΤΑ 1 στις χώρες του Νότου, που είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από αυτό το πρόβλημα και από τις συνέπειες της εξάπλωσης αυτού του ιού. Εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε και να παρακολουθούμε αδρανείς το θάνατο χιλιάδων πολιτών των χωρών αυτών του Νότου λόγω μιας πανδημίας ή λόγω ασθενειών που έχουν εξαλειφθεί μεν στις χώρες του Βορρά αλλά όχι στο Νότο. Ο Δάγκιος, η ελονοσία, η φυματίωση και όλα αυτά είναι πολύ μακρύς ο κατάλογος και παρόλα αυτά εμείς παραμένουμε αδρανείς και παρακολουθούμε με απάθεια αυτή την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να κάνουμε τι απαραίτητε προσπάθειε για να βελτιώσουμε την υγειονομική υπερίθαλψη όχι μόνο στι χώρες του, του Βορρά αλλά να δώσουμε και μια αποτελεσματική λύση στα προβλήματα των χωρών του Νότου. Θέλω να τονίσω μία ακόμα. Θέλω να θέσω ένα ακόμα ερώτημα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα με τη δράση των δημοσίων αρχών και μόνο για να μπορέσουμε να έχουμε μόνο από το δημόσιο τομέα την υποστήριξη πρέπει να δώσουμε ισότητα ευκαιριών σε όλες τις περιοχές του κόσμου και πρέπει να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών. Επίσης βρισκόμαστε εν αναμονή της, ε, ε, του εμβολιασμού στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες και ανησυχίες για τις παρενέργειες που μπορούν να προέλθουν από αυτά τα εμβόλια. Θα μπορέσουμε να δώσουμε τα απαραίτητα εμβόλια για τις χώρες του Νότου και θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν είναι ικανοποιημένη με το σύστημα με το οποίο αντιμετωπίζουμε ως μορφή πρόληψης μέσω της πρόληψης της πανδημίας, ενώ στο Νότο μόνο εκ των υστέρων αντιδρούμε. Οι ομιλητές τώρα που λαμβάνουν το λόγο προσωπικά. Ένα μισή λεπτό, ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνω το λαμβάνει το λόγο ο κύριο Σαλόμ και με μεγάλη συγκίνηση του δίνω το λόγο γιατί είναι παλιό μου συνάδελφο και σύντροφο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σα λόγια. Η τιμή είναι δική μου και να εργάζομαι σε αυτό το θεσμικό όργανο που εσείς είσαστε αντιπρόεδρος και προεδρεύετε σε αυτή τη συνεδρίαση για το ενδιαφέρον που προκαλεί αυτή η ερώτηση που δεν είναι άλλο παρά να υποστηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να προβλέπετε και να καταπολεμάτε η πανδημία της γρήπης H1N1 ή τα 1N1. Πέρα όμω από αυτό, για αυτή την πανδημία, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι νόσοι σήμερα πλήττουν άνισα τις χώρες, ε, τις ε, αναπτυγμένες χώρες σε σχέση με τις ε, μη αναπτυγμένες χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε με συγχωρείτε, στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε δεκάδες ε, χιλιάδες ε, ε, θύματα, πράγματα, πράγματα που αποφεύγουν οι ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε την υγεία των ανθρώπων αυτών. Αλλά δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι τα μέσα για να διασφαλιστούν. Για την καταπολέμηση του AIDS, της φημαστίωσης, της ελονοσίας κατά άλλων νόσων μολυσματικών. Χρειάζονται εμβόλια που σήμερα δεν έχουν στη διάθεσή τους και ούτε μπορούν να αγοράσουν. Απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παροτρύνω, όπω εκφράστηκε ο ε, Επίτροπο, να αναζητήσει συμμαχίε, να προωθηθούν προγράμματα, να ενεργοποιηθούν ε, οι χώρε χορηγοί, να υπάρξει ε, προσπάθεια ώστε οι αναπτυσσόμενε χώρε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε γενικά φάρμακα, σε προσιτέ τιμέ για του υπηκόου του. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ρέρο. Δεν δημιουργήθηκε, κανένα αίτημα δεν εκφράστηκε για τη διαδικασία Capture the για παρεμβάσεις ατομικές και θα λάβει τον λόγο ο Επίτροπος Ουρμπάνα για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Κύριε Όρμπαν, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πέρα από αυτά τα οποία ανέφερα στην έναρξη της παρέμβασής μου, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιες άλλες πτυχέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει διαρκώς και με και οικονομικά με υποστήριξη τα θέματα υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό με προγράμματα και σχέδια δημοσιονομικής αρρωγής και ενίσχυσης για τις εθνικές προτεραιότητες και την αρρωγή αυτή θα μελετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις εναλλακτικές λύσεις που σε σχέση με αυτά τα μέσα μπορούν να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των πανδημιών. Και όπως ε, ε, είχα αναφέρει ε, μέσα τώρα ρητά και κατηγορηματικά θα το πω δεν έχει τα τεχνικά και οικονομικά μέσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγοράσει αυτά τα εμβόλια αλλά ακόμα και έτσι συνεργαζόμενοι με τον ΠΟΗ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με διάφορες συμμαχίες και συνασπισμούς και συμφωνίες με τα ενδιαφερόμενα εμπλεκόμενα μέρη θα προετοιμάσουμε τις αναγκαίες απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε ως προς αυτά τα θέματα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με την παρέμβαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε η συζήτηση για αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ακριβώς δηλαδή την δήλωση της Επιτροπής για την χρηματοοικονομική και οικονομική κατάσταση στη δημοκρατία της Μολδόβας, της Μολδαβία. Και πάλι θα λάβει για άλλη μια φορά τον λόγο Επίτροπος Όρμπαν για να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση εξ ονόματος της Επιτροπής. Έχετε τον λόγο.